τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής ημέρας, καθώς επίσης και τα κείμενα έχουν δημοσιευθεί. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι. Εγκρίνονται λοιπόν τα χθεσινά συνοπτικά πρακτικά.